Θέλει κάποιο συνάδελφο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ζητήσω το λόγο στα πλαίσια του Catch αργότερα. Σήμερα το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι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 Σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούμε με την κοινή συζήτηση με τη δέσμη μέτρων του σιδηροδρόμου. Πρώτο ομιλητή στον Ιενό Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο, ο κύριο Ελκαντράουι. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα συζητούμε ένα πολύπλοκο θέμα και πολύ λεπτό. Αυτό του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο έχουν ήδη γίνει έντονες συζητήσεις και θα συνεχιστούν από ό,τι φαίνεται. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ του ανοίγματο αυτής της αγοράς, αλλά συνειδητοποιώ ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο, θα πρέπει να δούμε μεγάλη πρόσοχη ποιους ε, φορείς θέλουμε να έχουμε και υπό ποιες συνθήκες. Οι προτάσεις της Επιτροπής ε, είναι δεν είναι μυστικό για κανέναν, μη αποδεκτές, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν αρκετά υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την πυκνότητα, την δομή των ε, σιδηροδρομικών ε, ε, γραμμών και άλλα θέματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές που με βοήθησαν ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία δέσμη μέτρων πιο ισοσκελισμένη που θα ψηφιστεί αύριο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε το πακέτο αυτό, τη δέσμη αυτό, αυτήν σαν ένα μέσον που θα επιτρέπει να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και για να το επιτύχουμε θα πρέπει να έχουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ του ανοίγματο των ε, αγορών και της παροχής υπηρεσιών ποιότητας. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνονται επιλεκτικές επιλογές εκ μέρους κάποιων ε, ε, υπηρεσιών για τις πιο ελκυστικές γραμμές και να αφήνονται κατά μέρος οι λιγότερο ελκυστικές. Η δομή επίσης και θα πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ καλά και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τους διαχειριστές των υποδομών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά την, ε, τα εισιτήρια καθώς και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε σε μία δέσμη μέτρων που αποτελεί δεδομένου τη συμφώνηση η τριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Μεταφορών μία πολύ καλή βάση. Βεβαίως υπάρχει σχετική νομοθεσία για να μπορέσουμε να αντιταχθούμε στην επιλεκτική επιλογή. Οι διάφορες εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δουν ποια είναι, ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα Πώς προβλέπετε το άνοιγμα των αγορών και ίσως νέων φορέων εκμετάλλευσης και θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο αλλά βάση κανόνων. Η αγορά θα πρέπει να είναι δίκαια αν θέλετε και εδώ βεβαίως δεν είμαστε πάντα σύμφωνοι μεταξύ συναδέλφων για όλα. Κάποιοι συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες που κατά την άποψή μου αποδυναμώνουν αρκετά το κείμενο της Επιτροπής Μεταφορών και δεν είναι αποδεκτές. Όσον αφορά την ε, εργασία, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι συλλογικές συμβάσεις και ο κοινωνικός διάλογος να λειτουργεί. Όσον αφορά το θέμα των ε, εισιτηρίων επίσης θα πρέπει να το προσέξουμε. Νομίζω ότι έγιναν πολλά βήματα και κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει όσον αφορά το σύστημα των, ε, της παροχής των εισιτηρίων σε πολλές χώρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στον επόμενο ομιλητή θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Είναι στη διάθεσή μας τα πρακτικά πλέον. Υπάρχουν ενστάσεις δεν υπάρχουν. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Και τώρα δίνω το λόγο στον Ματιό Γκρός. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Α, διαδικαστικά ζητάτε το λόγο. Τι θέλετε. Προηγουμένως για τα πρακτικά ο Προεδρεύων